Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είπατε εκπρόσωπος και λυπούμε που απουσιάζει σήμερα. Σήμερα είναι σημαντική μέρα για την Ουκρανία. Η προετία, έχει την Προεδρία του ΑΣΕ για το 2013, κάτι που ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί. Είναι ένα προνόμιο, αλλά και ευθύνη, θα δώσει τη δυνατότητα στην Ουκρανία να ανταποκριθεί στο ύψος των προσδοκιών και των περιστάσεων, που σίγουρα οι προσδοκίες είναι υψηλές. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στις άλλες διμερείς σχέσεις, την περασμένη Δευτέρα έγινε στο Τάλ της ΕΣ Βρυξέλλες έγινε σύνοδος κορυφής με τη συμμετοχή του Προέδρου Γιαννούκοβιτς και του Προέδρου Βαν Ρόμποϊ και του Προέδρου Μπαρόσο. Η Κάτι Άστον ε, αναφέρθηκε στα διεθνή θέματα και ήμουν και εγώ παρόν ούτως ώστε να σε ενημερώσω όσον αφορά τις προοπτικές να υπάρξει μία σχέση βαθιών ε, εμπορικών σχέσεων στο εγγύς μέλλον και σε, με υψηλό επίπεδο προσδοκιών. Οι συζητήσει μα ήταν ειλικρινεί και έχω κάθε πεποίθηση ότι η Σύνοδος Κορυφής έθεσε επιτροχιά μια σχέση που θα πρέπει να είναι ευρύτερη και πιο συγκεκριμένη. Οι δύο βασικά αποτελέσματα της Σύνοδου Κορυφής είναι η οθέτηση του σχεδίου δράσεως που αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων και την υπογραφή του πρωτοκόλου για τη Συμφωνία Ατερικής Σχέσεως και Συνεργασίας που επιτρέπει στην Ουκρανία να συμμετέχει στα προγράμματα της Ένωση. Στην ημερήσια διάταξη επίσης η εσωτερική κατάσταση στην Ουκρανία, οι διαπραγματεύσεις που έχουν ξεκινήσει για τη Μελλοντική Συμφωνία Σύνδεσης και η διαδικασία της μεταρρύθμισης. Η Ουκρανία αποτελεί τμήμα των χωρών γειτονία. Προσπαθούμε λοιπόν να συσφίξουμε τις σχέσεις αυτές, τις γειτονικέ και με τη σειρά της είναι ένα κίνημα αν σκεφτείτε και την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ του Σαββατοκυριακού και τα συμπεράσματα των ημερών ε, διαπραγματεύσεων που έγιναν αυτή τη Δευτέρα που επέτρεψαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει τελικά ε, την ε, είσοδο της Ρωσίας στον ΠΟΕ. Τώρα σύνοδο κορυφής ερχόμαστε. Η κυβέρνηση ανέλαβε κάποιες σημαντικές υποχρεώσεις για μεταρρύθμιση οικονομική, κάτι που χαιρετίζουμε. Ε, πρόκειται πολλά πολλά για την μεταρρύθμιση του τομέα των ε, δημοσίων ε, προμηθειών που είναι κάτι σημαντικό για την καταπολέμηση της διαφθοράς συμφωνίας με το Εθνές Νομισματικό Ταμείο συνήφθηκαν και σημαντικές μεταρρυθμίσεις δρομολογήθηκαν στο βασικό ενεργειακό τομέα η Ουκρανική κυβέρνηση κατάφερε έτσι να σταθεροποιήσει την κατάσταση της χώρας σε σημαντικό βαθμό Προφανώς αυτό είναι σημαντικό, όμως ε, ανησυχούμε όσον αφορά τις ε, πολλές αναφορές που έχουμε για την επιδείνωση των, καταστάσεων της θεμελιώδης αγορές, ε, θεμελιώδη δικαιώματα στην Ουκρανία. ακούγονται καταγγελίες ανησυχητικές για την ελευθεροτυπία, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και την ελευθερία των, του συνεταιρίζεστε και το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ουκρανίας πρόσφατα ε, κατήργησε το Σύνταγμα του 2004 που υφετήθηκε κατά την ε, Πορτοκαλή Επανάσταση. Είναι λοιπόν το Σύνταγμα του 1996 που δίνει περισσότερες εξουσίες στον Πρόεδρο που τώρα έγινε, αυτό εφαρμόζεται τώρα πια, είναι μια απόφαση άκρος αμφιλεγόμενη και θα πρέπει μάλιστα η Ουκρανία να κάνει συνταγματικές μεταρρυθμίσεις ε, που θα είναι συμμετοχικές και ανοιχτές. Μια τέτοια διαδικασία θα πρέπει να έχει σαν στόχο τη δημιουργία ενός συστήματος βιώσιμου ισορροπιών όσον αφορά την εξουσία που να συνάδει με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Επίσης, ε, είναι ένα θέμα το οποίο αναφέρθηκε και στο δικό σας ψήφισμα του μηνός Φεβρουαρίου. Μια άλλη απόφαση πολύ πρόσφατα του Συνταγματικού Δικαστηρίου ε, που μπορεί να ερμηνευτεί τρόπος αφορά τη διάρκεια της θητείας του ε, παρόντος κοινοβουλίου. Ενώ το Σύνταγμα του 1996, το οποίο τώρα ισχύει, προβλέπει μια θητεία τετραετή, το Συνταγματικό Δικαστήριο αποφάσισε ότι η εξουσία του Κοινοβουλίου θα εκπνεύσει μετά από πέντε χρόνια μόνο, διότι εξελέγει κατά τη διάρκεια της περίοδου του Συντάγματος του 2004. Αυτή η απόφαση ε, δείχνει την προσέγγιση που ακολουθείται όσον αφορά την παρούσα κυβέρνηση. Για μία ακόμη φορά η Ουκρανία χρειάζεται πάρα πολύ μια διαδικασία συνταγματικής μεταρρύθμισης που θα είναι ανοιχτή και συμμετοχική αντί αποφάσεις που λαμβάνονται ε, βάσει των διαφόρων περιστάσεων. Τα τελευταία χρόνια το επίπεδο των πολιτικών ελευθεριών ήταν πολύ υψηλό στην Ουκρανία. Μία μετά τις άλλες οι εκλογές αναγνωριζόταν από αξιόπιστους θεσμούς και θεωρείται ότι πληρούσαν τις διεθνείς προδιαγραφές. Είναι λοιπόν λυπηρό να διαπιστώνουμε ότι οι τελευταίες δημοτικές εκλογές 31 Οκτωβρίου επεκρίθησαν από τους περισσότερους ε, παρατηρητές. Ακόμα και αν αυτές οι επικρίσεις ε, δεν αφορούσαν παρά μόνο τεχνικές και δικαστικές στοιχές, παρόλα αυτά είναι ένα βήμα πιστοχώρησης. Οι αξίες και οι αρχές της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι αρχές θεμελιώδης για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρχές επί των οποίων κάθε συμβιβασμός αποκλείεται έτσι δε περαιτέρω με έναν εταίρο βασικό όπως είναι η Ουκρανία. Είναι κοινέ οι αξίες για ένα κοινό μέλλον αυτές. Αυτή είναι η πρόκληση της σύνδεσης της σχέσης της μελλοντική μεταξύ της Ουκρανίας και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως όπως το κάναμε κατά τη διάρκεια κορυφής της περασμένης Δευτέρας και όσο υπάρχουν τα προβλήματα, θα πρέπει να συνεχίσουμε να στέλνουμε μηνύματα σαφέστατα όσον αφορά το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε Πεντεχούχτ. ο συνάδελφός ο κύριος Μπρόκ έχει τώρα το λόγο ως πρώτος ομιλητής από τα πολιτικά κόμματα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την δήλωση που έδωσε ο κύριος Ντεχούχ, εξ ονόματος της ΥΠΑ του εκπροσώπου, δεν έχω πολλά να προσθέσω. Νομίζω όμως ότι λόγω αιτίων που πρέπει να έχουν να κάνουν και με την κοινοβουλευτική σταθερότητα στην Ουκρανία έχει αποφασιστεί μια σειρά από μεταρρυθμίσεις. Ε, αυτό είναι πολύ θετικό. Οι τελευταίες βουλευτικές εκλογές ήταν ε, απόλυτα καθαρές, αλλά αυτό δεν συμβαίνει με τις δημοτικές εκλογές όπου υπήρξαν πολλές κατηγορίες και καταγγελίες από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλιστεί ότι οι δικαστικές εξουσίες θα αναλάβουν το καθήκον, το, το, το εκλογικό δικαστήριο, να εξασφαλίσει την αμεροληψία των εκλογών. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με τις κοινέ μας αξίες και έχει ένα αποφασιστικό ρόλο. Εφόσον λοιπόν μιλάμε για την ε, ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εξάλλου όμως είμαι ικανοποιημένο που τη Δευτέρα έγινε πρόοδο σε πολύ σημαντικά θέματα. Επομένως, δεν πρέπει αυτά τα οποία λέω από άποψη επικρίσεων να εμποδίσουν την πρόοδο στα θέματα της χωρίσης προξενικών θεωρήσεων και επίσης το θέμα της εμβάθυνσης των εμπορικών σχέσεων με την Ουκρανία και της ανάπτυξης μιας ζώνης πιο στενών εμπορικών σχέσεων. Αυτό θα οδηγήσει την Ουκρανία να έρθει πολύ πιο κοντά στην ευρωπαϊκή Ενία αγορά και αυτό σημαίνει ότι όχι μοναχά σε πολιτικό επίπεδο αλλά και σε οικονομικό επίπεδο η Ουκρανία θα πρέπει να γνωρίζει ότι το μέλλον της βρίσκεται στην Ευρώπη. Και η ευρωπαϊκή αγορά ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τις πρώτες ύλες τις οποίες μπορεί να παράσχει η Ουκρανία. <clears throat> Πιστεύω όμως κυρίες και κύριοι ότι θα πρέπει να είναι σαφές σε όλους μας ότι όχι μονάχα στο, με το συμφέρον, προς το συμφέρον της, Ουκρανίας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να εξασφαλίσουμε την ε, προσέγγιση μας με την Ουκρανία εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα με την Τουρκία και την προσέγγιση της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ από την ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και ο Σεβερίν έχει το λόγο θα μπορούσα να εκφράσω ως εξής τη θέση της ομάδας μου. Μη ζη... Ε, ρωτάτε τι μπορεί να κάνει η Ουκρανία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, <laughs> ρωτήστε τι μπορεί να κάνει... Μη ρωτάτε, συγγνώμη, τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ουκρανία. Το αντίστροφο ρωτήστε, παραφράζοντας το γνωστό απόφθεγμα. Ε, θα πρέπει να βασιζόμαστε σε δεδομένα και σε μια συγκεκριμένη στρατηγική στις σχέσεις μας με την Ουκρανία και νομίζω ότι πληρούνται τα κριτήρια ε, και ε, αυτό φάνηκε στην τελευταία σύνοδο και θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου προς τον Επίτροπο ε, θα θέλαμε να προσφέρουμε αρρωγή ε, προς την Ουκρανία και ε, υπάρχουν πολιτικές ε, ρήξεις στην Ουκρανία και δεν έχει σχέση όμως εμείς δεν πρέπει να τοποθετούμαστε ανάλογα με την, τον προσανατολισμό των διαφόρων κομματικών παρατάξεων δεν πρέπει να βασιζόμαστε σε φήμες θα χρειαζόμαστε πολιτικές ούτως ώστε η Ουκρανία να μπορέσει οργανικούς πώς να εισαχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι να χρησιμοποιήσουμε την Ουκρανία για να επιταχθούμε στις ε, γειτονικές της ε, χώρες. Ε, δεν είναι τέλειο το σημερινό ψήφισμα, αλλά είναι ένα καλό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης που προκρίνω και εγώ. Υπάρχουν κάποια λάθη μέσα στο ψήφισμα. Θα πρέπει να ζητήσουμε από όλους τους πολιτικούς φορείς της Ουκρανίας να αποφύγουν να το προβάλλουν ως μια νίκη εναντίον των άλλων. Δεν είναι αυτός ο στόχος του ψηφίσματος. Ο στόχος είναι όλες οι πολιτικές δυνάμεις της Ουκρανίας να πάρουν το μήνυμα ότι ήρθε η στιγμή να συσπηρωθούν πίσω από κάποιου κάποιους ελάχιστους στόχους για να έχουν αποτελέσματα και να εφαρμόσουν πολιτικές που θα επιτρέψουν στους πολίτες να ζουν καλύτερα και θα δώσουν μια καλύτερη ευκαιρία στην Ουκρανία να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν χρειάζεται να διεθνοποιούμε τις εσωτερικές συγκρούσεις της Ουκρανίας. Ε, ας εκπληρώσουμε εμείς τα καθήκοντά μας και θα ανταμυφθούμε από, το, από τις ίδιες μελλοντικές εξελίξεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε συνάδελφε Σεβερίν από πλευρά των φιλελευθέρων. Ε, κυρία Βαλέαν. Yes, thank Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Κύριε Επίτροπε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το να δούμε ότι η Ουκρανία τίθεται τόσο συχνά στην μέση διαταξή μας, αυτό αντικατοπτρίζει την πρόοδο στη σχέση μας. Εγώ πιστεύω ότι ο πραγματισμός, η πραγματιστική προσέγγιση και ο σεβασμός ο αμοιβαίος, η αναγνώριση των διαφορών αλλά και του κοινού συμφέροντος και η δημιουργία κοινών εγχειρημάτων και μιας εταιρική σχέσης είναι πολύ θετικά στοιχεία. Χαιρετίζω την δήλωση της Ουκρανικής ηγεσία που κατασυχάζουν ορισμένου φόβου ότι η Ουκρανία απέχει πολύ από την, το να γίνει μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά υπάρχει και μια διαμάχη μεταξύ ευρωπαϊκών ε, πολιτικών οικογενειών μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης στην, Ουγγαρία, στην Ουκρανία. Αυτό δεν βοηθάει. Αυτό δεν θα βελτιώσει ούτε τη θέση της κυβέρνησης, ούτε τη θέση της αντιπολίτευσης. Δεν είναι ένας ανταγωνισμός ποιο θα έχει την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να έχουν την υποστήριξη των ίδιων των πολιτών τους και να είναι μια δημοκρατία και ευμαρής χώρα η Ουκρανία. <clears throat> η διάσκεψη κορυφή η πρόσφατη έχει βοηθήσει πολύ το να υπάρξει καλύτερη πρόσβαση τη Ουκρανία στα ευρωπαϊκά προγράμματα και αναμένω ακόμα να υπάρξει μεγαλύτερη ε, προσέγγιση <clears throat> σε ε, μια σειρά από χώρους και επίσης τις θεσμικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει στον τομέα των μεταρρυθμίσεων πρέπει να εδραιωθούν περισσότερο. Ο νόμος περί δημοσίων προμηθειών ενεκρίθη στην αρχή του χρόνου, επομένω αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία παρέκκληση ακόμα και για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ε, Ποδοσφαίρου. Θα πρέπει επίση να βελτιωθεί το φορολογικό πλαίσιο, το οποίο δεν πρέπει να είναι άχθος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές για μια εύρωστη οικονομία. <clears throat> δεν πρόκειται όμως εμείς να πούμε στην Ουκρανία τι θα κάνει. Η Ουκρανία δεν πρέπει να κάνει πράγματα για μας, θα πρέπει η Ουκρανία να, να πράξει αυτά που είναι απαραίτητα για την δική της πρόοδο. Και οι πολιτικές και οι οικονομικές λοιπόν μεταρρυθμίσεις είναι προϋπόθεση για ένα καλό μέλλον για την Ουκρανία που θα είναι προ το καλύτερο συμφέρον των πολιτών τη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Βαλεάν <clears throat> για τους πράσινους Ελεύθερη Ευρωπαϊκή Συμμαχία η κυρία Χάμς για δύο και μισά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είδαμε στις τελευταίες μέρες στο Χακίβ, στο Λουγκάν, στο Κίεφο και σε άλλες μεγάλες και μικρές πόλεις στην ε, Ουκρανία είδαμε να γίνονται μεγάλες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας. Δεκάδες, εκατοντάδες μέχρι χιλιάδες πολιτών της Ουκρανίας κατέβηκαν στους δρόμους. <clears throat> Διαμαρτύρονται για το φορολογικό καθεστώς το οποίο θεωρούν ότι είναι άδικο και αν πρέπει το ψήφισμά μας να κατευθυνθεί σε κάποιους εγώ νομίζω ότι θα πρέπει κατά κύριο λόγο να απευθύνεται στους πολίτες της Ουκρανίας που με τις διαμαρτυρίες τους εξασφαλίζουν ότι πράγματι θα προχωρήσει η δημοκρατική μεταρρύθμιση στην Ουκρανία. <clears throat> Το ψήφισμά μας, το οποίο εκφράζει φόβους για μια διάβρωση της δημοκρατίας στην Ουκρανία, φυσικά συνδέεται άμεσα με αυτές τις ε, διαδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά της κυβέρνησης και του κρατου, κρατικού μηχανισμού στην Ουκρανία. Αυτές λοιπόν οι διαδηλώσεις ε, προβλέπεται να λάβουν χώρα και αύριο. Πρόκειται για εκατοντάδες χιλιάδες ίσως και μέχρι ένα εκατομμύριο στο Κίεβο που θα κατέβουν στον δρόμο. Όλα αυτά με μεγάλο ενδιαφέρον τα παρακολουθώ, αλλά όχι και χωρίς κάποιες ανησυχίες σε σχέση με αυτή την εξέλιξη. Έχει δείξει η κυβέρνηση της Ουκρανίας ότι μέχρι σήμερα ξεκολουθεί να υπάρχει ελευθερία του Συνέρχεστε, Ελπίζω ότι θα συνεχίσει να το πράττει αυτό. Το ψήφισμά μας έχει γίνει με τη συμμετοχή πολλών πολιτικών ομάδων. Νομίζω θα ήταν λαθασμένο για την εξέλιξη της Ουκρανίας αν εμείς μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρχίσουμε να διχαζόμαστε μεταξύ των κομμάτων που υποστηρίζουν τη συμπολίτευση στην ε, <clears throat> Ουκρανία και άλλοι να υποστηρίζουν την κυρία Τιμοσέγκο. Αυτά δεν πρόκειται να βοηθήσουν την εξέλιξη της δημοκρατίας στην, Ουγγαρία, στην Ουκρανία. Συγγνώμη. Επίσης πιστεύω ότι το ψήφισμα αυτό το οποίο έρχεται αμέσως μετά την διάσκεψη κορυφής με την Ουκρανία, ακριβώς λόγω των μεγάλων διαδηλώσεων και των διαμαρτυριών και των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν για τις μεταρρυθμίσεις στην Ουκρανία, πρέπει το ψήφισμά μας να έχει ένα ιδιαίτερα εχμηρό χαρακτήρα και να αντιμετωπίσει τις διαμαρτυρίες και τις διαδηλώσεις που γίνονται. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την προσοχή σας και ελπίζω θα μπορέσουμε και μαζί με την Κομισιόν να βοηθήσουμε αυτή τη χώρα που είναι τόσο κοντά σε εμά τους Ευρωπαίους και να δείξουμε και την αλληλεγγύη μας προς την Ουκρανία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Χάμς, ακολουθεί για την ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών ο κύριος Κόβαλ. 1,5 λεπτό. E, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ πολλές εβδομάδες πέρασαν ήταν πολύ ενδιαφέρουσε συζητήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που αφορούσαν την Ουκρανία και το μέλλον της χώρας. Νομίζω ότι η Ουκρανία παρακολουθεί αυτά που λέμε εμείς και γι' αυτό θα πρέπει το ψήφισμά μας να το θεωρήσουμε ως επιστολή. Όχι ως επιστολή υπό συγκεκριμένο κόμμα, αλλά ως ένα μήνυμα προς τους Ουκρανούς. Μια επιστολή στην οποία θα μιλούμε με ενδιαφέρον θα μιλούμε ως γείτονες, οι οποίοι γείτονες είναι ανοιχτοί και θέλουν να αγκαλιάσουν τους Ουκρανούς. Ευχαριστώ πολύ τη Ρεμπέκα Χάρμς που ξέρει πολύ καλά τι να πει. Οι εκλογές δεν ήταν ικανοποιητικές, δεν ήταν ιδεώδεις οι συνθήκες, αλλά πρέπει να πούμε ότι υπάρχει κάποια ευκαιρία για την Ουκρανία και θέλουμε να την υποστηρίξουμε την Ουκρανία θα πρέπει να αναφερόμαστε στα θετικά στοιχεία επίσης. Μόνο στον οικονομικό τομέα έχουν συμβεί τα θετικά γεγονότα. Θα πρέπει να αναφέρουμε και τον πολιτικό τομέα όμως. Να δείξουμε ότι η πόρτα της Ευρώπης είναι ανοιχτή για την Ουκρανία και είναι καλό ότι αυτό ήταν το μήνυμα της Συνόδου Κορυφής και είναι πολύ καλό το ότι σήμερα λέμε ότι το ψήφισμα δεν αφορά συγκεκριμένο κόμμα, αφορά τους Ουκρανούς όλους και το υθετήσαμε όλοι μαζί. Σα ευχαριστώ κύριε Κόβαλ. Ακολουθεί για ένα λεπτό από την ομάδα της Νομόσπονδης Ευρωπαϊκής Αριστεράς, Βόρειας Καναδική Αριστερά, ο κ. Κόουλιτσεκ. Ευχαριστώ. Ε, ε, λοιπόν, είναι καλό το ότι συζητούμε το θέμα αυτό για την Ουκρανία. Ε, μας θυμίζει η όλη εικόνα τον κύριο Κρίτσικο, τον μποξέρ που είναι κάποιο άλλους μποξέρ. Ε, είναι επίσης βαρέων βαρών και η Ουκρανία σαν χώρα και πολλά ε, εξαρτώνται για τη διέλευση από κεντρική ε, Σιβηρία και από πιο μακριά που περνούν από την Ουκρανία. Η Ουκρανία είναι πάρα πολύ σημαντικό φορέα και γι' αυτό καλωσορίζω την συνεργασία που υπήρξε με τη Ρωσία και το αποτελέσμα τη Συνόδου Κορυφή Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Ε, είναι σημαντικό τμήμα του εργατικού δυναμικού στις περισσότερες ε, χώρες. Τα βασικά προβλήματα της χώρας αυτής μοιάζουν με πολλές, πολλά προβλήματα που έχουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ε, ανεργία, ε, προβλήματα στον φατιστορήσεις διαβατηρίων κλπ. Σύμφωνα στους παρατηρητές, οι εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση δεν δημιούργησαν προβλήματα. Το ψήφισμα που υπέβαλαν τα πολιτικά κόμματα είναι ένας καλός συμβιβασμός και θέλω να τον υποστηρίξω. Ευχαριστώ πολύ. Ακολουθεί για την ομάδα της Ευρώπης, της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας ο κ. Μπέλντερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. <clears throat> Πολλές φορές είναι εντυπωσιακές οι ελλείψεις κανονικότητας στις τοπικές και τις περιφερειακές εκλογές στην Ουκρανία θα πρέπει να είναι κόδωνας κινδύνου για την Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρξε μαζική νοθεία προσθήκη ψηφοδελτίων και σε ορισμένε περιπτώσεις φωτοτυπήθηκαν ορισμένα ψηφοδέλτια και υπήρξε πίεση σε πολλούς να μην κατέβουν σε εκλογές στα κόμματα τη αντιπολίτευση. Αυτό ήταν μια απόλυτα αντιδημοκρατική διαδικασία. Βέβαια, <clears throat> οι προηγούμενε κοινοβουλευτικέ εκλογέ ήταν καθαρέ, αλλά θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει στι εκλογέ του 2012 θα πρέπει να αναχαιτήσουμε τις αυταρχικές κινήσεις στην Ουκρανία γιατί εμπλέκεται και η δική μας αξιοπιστία έναντι των ελίτ της χώρας και των δημοκρατών που θέλουν μια μεταρρυθμίση στην Ουκρανία. Ελπίζω <clears throat> ότι ακόμα δεν έχουμε λόγους για σοβαρές ανησυχίες. <clears throat> Ευχαριστώ τον κύριο Μπέλντερ. Ακολουθούει ο κύριος Μέλτσερ για τους μη εγγεγραμμένους. <clears throat> Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ξέρουμε όλοι ότι η Ουκρανία είναι μία από τις πιο κοντινές γειτονικέ χώρες της Ευρώπης και ότι έχει μια πολύ μεγάλη δυναμικότητα για το μέλλον. <clears throat> Είναι επομένω ένα πολύ σημαντικό εταίρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν πρέπει από πολιτική άποψη να βρεθεί μακριά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά παρόλα αυτά είδαμε ότι κέρδισε η, στις τοπικές εκλογές η παράταξη που υποστηρίζει την ε, ρωσική επικυριαρχία ούτως Είναι σημαντικό λοιπόν οι Ευρωπαίοι να καταφέρουν να επιλέξουν οι Ουκρανοί τις ευρωπαϊκές αξίες, όχι τις αξίες κάποιων άλλων και όχι να υποκύψουν στα παιχνίδια της γειτονική υπερδύναμης. Θα πρέπει να τους θεωρήσουμε ότι είναι ίσοι εταίροι και εμείς και η Ρωσία εξάλλου. <clears throat> Ο στόχος μας δεν πρέπει να είναι κατά να υπάρξει ενσωμάτωση της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να κάνει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και μόνο τότε μπορεί να αποφασίσει αν θέλει να παραμείνει ανεξάρτητη και αυτόνομη ή να ενσωματωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριε Μέλτσερ. <clears throat> Ακολουθούν οι υπόλοιποι ομιλητές. Καταρχήν ο κύριος Γκάλερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. <clears throat> Πράγματι υπάρχει μεγάλη δυνατότητα συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ουκρανία και αυτό το κατέδειξε η διάσκεψη κορυφή το πρόγραμμα για την απελευθέρωση των προξενικών ε, θεωρήσεων και η σχετική συμφωνία είναι ένα δείγμα αυτή της δυνατότητας. Έχουμε υποστηρίξει όλο αυτό το συμβαστικό ε, ψήφισμα για να τονίσουμε ιδιαίτερα τα θετικά στοιχεία τα οποία μπορεί να έχει η συνεργασία μας με την ε, Ουκρανία. Αλλά όπως λένε οι Άγγλοι, the proof of the pudding is in the eating. Θα φανεί στην πράξη εάν μπορούμε πράγματι να υλοποιήσουμε όλο αυτό το δυναμικό που υπάρχει στη σχέση μας με την Ουκρανία. Ε, είναι ε, ήδη το θέμα αυτό των δημοσίων διαγωνισμών το οποίο ανέφερε ο κύριος ε, Επίτροπος και μεταξύ άλλων και οι διαγωνισμοί, οι προμήθειες για το Ευρωπαϊκό Ποδόσφαιρο, Ποδοσφαίρου που δεν καλύπτονται από τη νέα νομοθεσία. <clears throat> Αυτό θα πρέπει να μας οδηγήσει σε κάποιες ανησυχίες. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τον κύριο ε, επίτροπο, ο οποίο αναφέρθηκε για τι ανησυχίε που έχουν να κάνουν με τα μέσα ενημέρωση, το δικαίωμα συνέρχεστε κτλ. Και σίγουρα είναι ένα βήμα προ τα πίσω η κατάσταση που έλαβε χώρα στι εκλογέ. Εμεί θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό και το τονίσαμε πράγματι μέσα στο ψήφισμά μα. Για τον κύριο Σέβεριν, εγώ δεν νομίζω ότι πρέπει να διεθνοποιούμε τις εσωτερικές ε, διαμάχες μέσα στην Ουκρανία. Αυτό είναι μια αναδιατύπωση της βασικής αρχής της μη ανάμειξης στα εσωτερικά άλλων χωρών. Αυτή είναι η βασική μας αρχή. Δεν πρέπει λοιπόν ακριβώς με την Ουκρανία, επειδή θέλουμε να την ε, προσελκύσουμε στην Ευρώπη, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή τη χώρα με ευρωπαϊκά μέτρα και σταθμά και επομένω είναι πολύ σωστό, όπως είπε και η κυρία Χάμς, να συνεχίσουμε να έχουμε στενέ επαφέ με την Ουκρανία και να εξασφαλίσουμε ότι όταν πρόκειται για δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα δεν θα υπάρξουν οι παραχωρήσεις στην πολιτική γραμμή της. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γκάλου. Ο κύριος Φόμποντα, για ένα μισή λεπτό έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, <clears throat> δυστυχώς δεν έχει εκπληρώσει τις υποσχέσεις της η πορτοκαλή επανάσταση Βλέπουμε τι έχει γίνει μεταξύ Γιαννούκοβιτς και Τιμοσέγκο και Ιουσέγκο. Και επίσης οι δημοτικές εκλογές δεν επέτυχαν το στόχο τους, δεν μπόρεσαν να ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα για διαφάνεια. Και αυτό είναι φανερό λοιπόν στην Ουκρανία. Κύριε Γκάλερ, αυτό το οποίο είπε ο κύριος Σέβεριν λέει ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε μια σαφή γλώσσα και έναντι της κυρίας Τιμοσέκο. Να πούμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να έρθει προς την κατεύθυνση Ευρώπη Ευρώπης και να αφήσει κατά μέρο τους ολιγαρχείς στη χώρα αυτή. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι εμεί θέλουμε να διαταράξουμε την κοινοβουλευτική διαδικασία στην Ουκρανία. Πράγματι θέλουμε να διατηρηθούν τα ευρωπαϊκά δημοκρατικά πρότυπα. η πράσινη δεν είναι πάντα στη μέση ανάμεσά μας, αλλά ίσως μπορούμε να ακούσουμε αυτή τη φορά αυτά που είπε η κυρία Χάρμς. Ας βοηθήσουμε τη χώρα αυτή να προοδεύσει και να ακολουθεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τα, την ευρωπαϊκή ιδέα για την ένωμη τάξη. Αυτή είναι η πολιτική που ακολουθούμε λοιπόν εμείς. Και το κάνουμε αυτό χωρίς ιστεροβουλία. Έχουμε επικρίνει μεν αυτά τα οποία έγιναν στις εκλογές, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει κύριε Μπρόκ να είναι επικοδομητική <clears throat> η αντιπολίτευση και εσείς ήταν επικοδομητικός τόσες πολλές φορές. Επομένως πείστε την κυρία Τιμοσέγκο να κάνει αυτά που έκανε και ο κύριος Γιανακόβης. Ευχαριστώ κύριε Σφόμποντα. Ακολουθεί ο κύριος Μιγκάσκι για ένα μισή λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ξεκινήσω με αυτά που είπε και ο Σεβερίν, που είπε κάτι σημαντικό Δηλαδή θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για την Ουκρανία και όχι τι μπορεί να κάνει η Ουκρανία για μας. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σεβερίν για αυτά τα λόγια, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας. Οι εκλογές δεν πήγαν πολύ καλά. Σύμφωνα με τις δικές μας προδιαγραφές και πρότυπα υπήρξαν ε, ε, κάποια προβλήματα, αλλά δίκιο έχει η κυρία Χάνς, η οποία είπε ότι η δουλειά μας δεν είναι να κοιτάμε προς τα πίσω, αλλά ε, να μην κοιτάμε τι κάνει το ένα το άλλο κόμμα, τι κάνουν οι Ουκρανοί και τι θέλουμε εμείς, διότι η ένταξη της Ουκρανίας είναι προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και προς όφελος και των Ουκρανών. Και νομίζω ότι το να προχωρούμε πολύ μακριά και να θέλουμε πολλά από τους Ουκρανούς δεν είναι κάτι ειλικρινές, διότι εδώ, σε αυτή την αίθουσα, υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι είναι πολύ φιλελεύθερη όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και για άλλα ζητήματα για, όσον αφορά τους εταίρους τους, αλλά είναι πολύ απαιτητική έναντι της Ουκρανίας. Και αξίζουν την υποστήριξή μας οι Ουκρανοί, ανεξάρτητα από το πολιτικό κόμμα προς το οποίο απευθυνόμαστε και που συζητούμε. Και να θυμάστε ότι αυτό που διακυβεύεται εδώ είναι η πιο στενή επαφή μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ενώσης και της Ουκρανίας. Ευχαριστώ κύριε Μιχάλσκι. Ο κύριος Κάμπελ Μπάνγκημαν έχει το λόγο. Για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, ξέρω την Ουκρανία από επισκέψεις στο Κίεβο και στην Κρυμαία και συλλέγονται Τέκο και Τσίσκο, Ουκρανού καλλιτέχνε. Οι Ουκρανοί είναι καλοί, ε, θερμοί, γενναιόδοροι άνθρωποι, αλλά πολιτικό σκοπό θα πρέπει να προσέξουμε πολύ. Η Ουκρανία είναι μια χώρα που είναι διρεμένη μεταξύ δυτικών που είναι υπέρ τη Δύσεω, τη Δύση που είναι υπέρ τη Δύσεω και τη Ανατολή που είναι υπέρ τη Ανατολή και τη Ρωσία. 45 εκατομμύρια πολίτε έχει και η Ρωσία θεωρεί ότι είναι στην αυλή τη αυτή η χώρα. Ε, υπάρχει ο ρωσικός στόλος στη Σεβαστόπολη ε, και θα διαφυλάξουν αυτή την πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα από εκεί οι Ρώσοι και οποιοδήποτε αίτημα για την Ουκρανία να μπει ε, στο ΝΑΤΟ θα είναι κλωτσιά προς τη ρωσική αρκούδα. Λοιπόν, δεν θέλουμε να αυξήσουμε τις εντάσεις σε δύσκολους καιρούς και το να πιέσουμε την Ουκρανία από επιδοτήσεις αγροτικές κλπ να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το κόστο θα είναι απαγορευτικό. Να τη βοηθήσουμε καλύτερα με άλλο τρόπο και να αφήσουμε την Ουκρανία σαν μια υπερήφανη ανεξάρτητη χώρα που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κάμπελ Μπάνεμαν. Η κυρία Σέιντι έχει το λόγο. Ο κύριο Σέιντι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Νομίζω μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε πως ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω ε, πληθυσμού ε, και λόγω γεωγραφικής θέσης η Ουκρανία είναι βασικός γεωστρατηγικός εταίρος. Αλλά λείπουν δύο πράγματα μέσα στο ψήφισμα. Δεν αναφερόμαστε καθόλου στις εθνικές μειονότητες 65% του πληθυσμού είναι Ουκρανοί και μετά έχουμε διάφορες εθνικότητες, Ούγγρους, Ρώσους, ε, Τατάρους, Ρουμάνους ε, ε, που ζουν στην Ουκρανία. Θα θέλαμε το ψήφισμα αυτό να συμπεριλαμβάνει και τα αιτήματά μας σχετικά με τις μειονότητες, δηλαδή να κατοχυρωθεί η παιδεία σε γλώσσες των μειονοτήτων, Επίσης, ε, να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ε, προστασίας της πολιτιστικής ε, κληρονομιάς, όπου στην περιοχή πέρα από τα Καρπάδια όπου καταστράφηκαν μοναστήρια και για τις εκλογές θα έπρεπε να διευκρινίσει τη θέση της Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε. Ο συνάδελφος Σαλεύσκη τώρα. E, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. <clears throat> Ήταν μια πάρα πολύ σημαντική εβδομάδα για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουκρανίας. Ήταν μια πάρα πολύ επικοδομητική εβδομάδα από αυτή την άποψη. Καταρχήν τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια της διάσκεψης κορυφής, δημιουργήσαμε από κοινού ένα οδικό χάρτη ο οποίος ε, θα προωθήσει τη φιλελευθερωποίηση του καθεστώτος προξενικών θεωρήσεων. Και εξάλλου, αύριο θα ψηφίσουμε ένα ψήφισμα το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ θετικό από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο θα διανοίξει το δρόμο σε περαιτέρω συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανίας. <clears throat> Δίνει αυτές τις δυνατότητες λοιπόν και στις δύο πλευρές και περατώνει τις συζητήσεις οι οποίες θα έχουν λάβει χώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι έχουμε καταλήξει σε μια συμβαστική λύση και έχουμε μια ενιαία και κοινή θέση. Δεν απευθυνόμαστε μόναχα σε μεμονωμένες ομάδες και πολιτικά κόμματα στην Ουκρανία, στο κόμμα του κ. Γιάννου Κοβετσίτη, κ αλλά σε όλο το Ουκρανικό έθνος τους παρακινούμε να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις ώστε να εξασφαλίσουν τη μελλοντική τους ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι σημαντικό επίσης να αξιολογήσουμε τη λειτουργία της κυβέρνησης και του διοικητικού μηχανισμού στην Ουκρανία βάσει των πραγματικών τους επιτευγμάτων. Αυτή είναι και η πρώτη κυβέρνηση, σας υπενθυμίζω, που έχει εφαρμόσει ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων συνεργαζόμενοι με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και θεωρούμε ότι έχουν δρέψει τους καρπούς αυτής της προσπάθειας στην οικονομία. Η κατάσταση αδιεξόδου σε πολιτικό επίπεδο που έχει λάβει χώρα στην Ουκρανία τα τελευταία χρόνια μπορεί, είναι σε ένα σημείο που μπορεί πράγματι να τερματιστεί. Και πρέπει η Ουκρανία να προχωρήσει στον δρόμο των φιλοδοξιών της να γίνει τμήμα της Ευρώπης. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε αυστηροί με αυτά που έγιναν στι εκλογέ. Ευχαριστώ κύριε Ζαλεύσκη. Ο κύριο Σίβιετ, για ένα μισή λεπτό. Σήμερα συζητούμε σε ένα διαφορετικό κλίμα δεν υπάρχουν πια συναισθηματισμοί και η διατύπωση στο ψήφισμα απηχεί καλύτερα την πραγματικότητα. Είναι πάρα πολύ καλό. Προσπαθούμε με ενιαία φωνή να εκφραστούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρά τις δυσκολίες που έχουμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν. Εδώ δεν μιλάμε για την ποιότητα της δημοκρατίας στην Ουκρανία. Συζητούμε για την αποτίμηση της ποιότητας ε, της δημοκρατίας, ε, τον τρόπο αποτίμησης. Έχουμε τους, ε, ε, τις διάφορες επαναστάσεις, ε, τις διάφορες πολιτικές παρατάξεις, η μπλε, η πορτοκαλί, μετά πάλι η μπλε, μετά πάλι η πορτοκαλί ο κύριος Γιαννούκοβιτς και όλα τα κόμματα της Ουκρανίας θα πρέπει να πάρουν το μήνυμα ότι πρέπει να επομιστούν την ευθύνη για την προστασία Τη κληρονομιά και για τα γεγονότα που ε, σημειώθηκαν πριν από λίγα χρόνια. Η Γιούλια Τιμοσέγκο θα πρέπει να ακούσει αυτό το μήνυμα γιατί είναι υπεύθυνη για την εικόνα τη αξιωματική αντιπολίτευση. και πρέπει να κατανοήσει ότι το να εκπροσωπεί την αξιωματική αντιπολίτευση δεν σημαίνει ότι απλώ θα κρατά την εξουσία. Πρέπει, οφείλει να εισηγηθεί μια εναλλακτική λύση που θα υιοθετήσουν ενδεχομένω ε, οι πολίτε ε, τη Ουκρανία διότι οι πολίτες ε, αντιλαμβάνονται την κατάσταση και έτσι μόνο θα στεφθεί με επιτυχία το εγχείρημά μας. Ε, ε, επειδή τους υποστηρίξαμε Ο, ο Κρίτσκο είναι πολύ γνωστός μποξέρ από την Ουκρανία, αλλά δεν υπάρχει μόνο αυτός. Ε, ευχαριστούμε κύριος Κίλαμ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα της καταρρεύσεως Σοβιετικής Ενώσεως ήταν η δημιουργία ανεξάρτητης Ουκρανίας. Είναι μια χώρα που θεωρείται σαν μελλοντικό μέλος της ευρωπαϊκής κοινότητας δεν μπορώ παρά να καλωσορίσω το ότι ο πρόεδρος Γιαννουκόβιτς και το νέο κοινοβούλιο επιβεβαίωσαν αυτές τις προσδοκίες για την προσχώρηση στην Ευρώπη. Διότι πραγματικά ανεξάρτητη και δημοκρατική Ουκρανία που είναι άνευ διαφθοράς και δεν θα φοβάται τους σωματοφύλακες και την μεγάλη σημαντική εξουσία, μια Ουκρανία με κράτος δικαίου θα είναι ένας παράγοντας σταθερότητας για όλη την Ήπειρο. Χωρίς πραγματική δημοκρατική Ουκρανία δύσκολα φανταστεί κανείς πραγματικά δημοκρατική Ρωσία. Χθες πέρασαν έξι χρόνια από την αρχή της Πορτοκαλή Επαναστάσεως. Δυστυχώς το τεράστιο δυναμικό αυτής της αλλαγής ε, σπαταλήθηκε. Όμως, χάρη στη νίκη των δημοκρατικών ε, διαδηλωτών το Δεκεμβρίου 2004 η αξιοπιστία των πολυκομματικών εκλογών και η ελευθεροτυπία ε, επεκράτησαν. Στο σχέδιο ψηφίσματο του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει ανησυχία όσον αφορά τον αυξανόμενο αριθμό αναφορών ότι οι δημοκρατικές ελευθερίες και τα δικαιώματα όπω είναι τα ελεύθερα μέσα ενημέρωση, ε, τελούν υπό απειλή και ότι οι υπηρεσίε ασφαλεία ξανάρχισαν να παρεμβαίνουν στις δημοκρατικέ δραστηριότητε των πολιτών. Ένα σημαντικό μήνυμα προς τη νέα κυβέρνηση είναι το εξής. Η Ευρώπη είναι ανοιχτή για όλους τους τομείς συνεργασίας. Το τίμημα συνεργασίας δεν είναι τίποτα λιγότερο από την αποκατάσταση των πλήρων ελευθεριών. Σαν πραγματικοί φίλοι της Ουκρανίας πρέπει να είμαστε φιλικοί και συνεπείς προωθώντας τις αξίες μας. Είναι λυπηρό το ότι έξι χρόνια αργότερα η νέα Ελίτεξ ακόμα δεν μπορεί να δεχτεί ότι η Πορτοκαλή Επανάσταση ήταν πραγματική έκφραση της λαϊκής βούλησης. Για να αντιμετωπιστούν τα αποτελέσματα τα, όταν καταλάβουν τα αποτελέσματα αυτής της, και τα κίνητα αυτής της επαναστάσεως που θα ολοκληρωθεί καλύτερα η κοινωνία της Ουκρανίας. Ευχαριστώ. Ακολουθεί η κυρία Κολάρσκα Μπομπίνσκα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε δεν θα αναφερθώ στο τι θα κάνουμε εμείς για την Ουκρανία ή τι πρέπει να κάνει η Ουκρανία για μας. Θέλω να μιλήσω σχετικά με τι θα πρέπει να κάνει τον εαυτό της Ουκρανία, η Ουκρανία ή την Ουκρανία. Η Ουκρανία θέλει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ακούμε και αναφορές για παραβιάση των θεμελιωδών ελευθεριών. Τις πρόσφατες μέρες ακούσαμε από δημοσιογράφους του PFI του τηλεοπτικού σταθμού που μας μίλησαν, που αναφέρθηκαν μάλλον, σε παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους και έχουμε πληροφορίες από ανεξάρτητες ε, πηγές ότι από 65 μεταρρυθμίσεις που είχαν προγραμματιστεί μόνο 4 πραγματοποιήθηκαν και σε πρόσφατη συζήτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάποιοι θεώρησαν ότι αν κατηγορήσουμε, καταγγείλουμε τις ατασταλίες και τις παρατυπίες θα αποθαρρύνουμε την Ουκρανία από τον ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι είναι καλύτερο να μην την επικρίνουμε την Ουκρανία και μόνο να την ενθαρρύνουμε για να πραγματοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις. Εγώ τι πιστεύω. Πιστεύω ότι καταρχάς πρέπει να προστατεύσουμε τις δημοκρατικές αξίες. Θα πρέπει να μιλάμε για αξίες και η κυβέρνηση θα πρέπει να μιλά για τις μεταρρυθμίσεις. Εμείς θα πρέπει να κατηγορούμε και να καταγγέλουμε τις παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων θα πρέπει να παράσχουμε μέσα για την πρόθεση της δημοκρατίας. Και χαίρομαι που υπογράψαμε ένα πρωτόκολλο σύμφωνα με το οποίο η Ουκρανία θα έχει πρόσβαση σε κάποια από τα προγράμματά μας και θα έχει επικρατήσει και καθεστώς απελευθερωμένο όσον αφορά τις θεωρίες διαβατηρίων. Αλλά η Ουκρανία πρέπει να κάνει μεταρρυθμίσεις. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κολάρσκα. Περνάμε τώρα στην οφθαλμοθυρευτική διαδικασία. Ο κύριος <laughs> Σφόμποντα έχει ήδη κάνει πολλές τέτοιες παρεμβάσεις αυτού του είδους. Είναι ίσως λιγότερες παρεμβάσεις από ό,τι φοβόμαστε στην αρχή, αλλά περισσότερες από ό,τι μπορούμε να αποδεχτούμε. Δίνω λοιπόν τον λόγο στον κύριο Κοσλόφσκι πρώτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, στην Ολομέλεια του Οκτώβρη ε, τόνισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα πρέπει να εξετάζουμε τη σχέση με την Ουκρανία από τρεις πλευρές. Ε, υπάρχει ε, διπουργική διάσκεψη ή ε, τοπικές εκλογές και η Σύνοδος Κορυφής. Εγώ με τον κύριο Κάβαλ παρακολουθήσαμε τις εκλογές. Δυστυχώς σημειώθηκαν αλλαγές στον εκλογικό νόμο τρεις μήνες πριν από τις εκλογές. Το Σύνταγμα του 2004 προβλέπει ότι Χρειάζεται σταθερότητα δικαίου, αλλά στην Ουκρανία δεν υπάρχει αυτό. Σημειώθηκαν επίση παρατυπίε και νοθεία στι εκλογέ και υπάρχουν αμφιβολίε για τα δημοκρατικά πρότυπα. Επίση, είναι επιτακτική ανάγκη να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά και να αναβαθμίσουμε τη δημόσια διοίκηση. Ελπίζουμε ότι με αυτό το ψήφισμα η Ουκρανία θα βοηθηθεί για να ακολουθήσει τον οδό των οικονομικών και πολιτικών μεταρρυθμίσεων. Ευχαριστούμε η κυρία Πίνκε Βιτσιούτε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι γεγονός ότι το συμβαστικό ψήφισμα για την Ουκρανία επέχει δική σημασία τόσο για τους λαούς, τον λαό της Ουκρανίας αλλά και για τους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι η Ουκρανία είναι ένας πολύ σημαντικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιδίως μέσα στα πλαίσια της πολιτικής γειτονίας. Είναι σημαντικό λοιπόν να προωθήσουμε αυτή τη συνεργασία ιδιαίτερα στο, στο καθεστώς προξενικών θεωρήσεων. Επομένως, η Κομισιόν θα πρέπει να προωθήσει την φιλελευθερωποίηση αυτού του καθεστώτος όσο το δυνατόν συντομότερα. <clears throat> Επίσης, για τη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου θα πρέπει να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε την σταθερότητα στα όμορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συνταγματικέ μεταρρυθμίσεις μεν έχουν μεγάλη σημασία, πρέπει να κατανοήσουμε όμως ότι χρειάζεται χρόνος για να επιτευχθούν και επομένω δεν θα πρέπει μόνο να επικρίνουμε, θα πρέπει να βοηθούμε και την Ουκρανία να ενσωματωθεί στην ευρωπαϊκή μα οικογένεια. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πίνκε Βιτσιούτε. Η κυρία Οβίερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Επίτροπε, συνάδελφοι. Μπορούμε ε, να πούμε ότι τίποτα δεν είναι προβλέψιμο στην Ουκρανία. Χαίρομαι πάρα πολύ όμως που αυτό ο ισχυρισμό δεν ισχύει πια γιατί η κυβέρνηση κατάφερε να σταθεροποιήσει την κατάσταση και ανθεί η οικονομία η Ουκρανία. Ενδιαφέρεται για τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά είναι αμφίδρομο αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ενδιαφέρεται να ε, υπάρχει, υπάρχουν κράτη δικαίου ε, πέρα από τα σύνορά της. Υπάρχουν βέβαια προβλήματα σε σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ουκρανία, αλλά Σίγουρα δεν θα υποχωρήσουμε ως προς τα αιτήματά μας και χρειάζεται να συνεργαστούμε με την Ουκρανία. Πρέπει να πούμε επίσης ότι η απόφαση που ελήφθη πριν από ένα μήνα εδώ στο Κοινοβούλιο για την αναβολή της ψηφοφορίας αυτής, αυτού του ψηφίσματος ήταν σοφή. Αύριο θα εγκρίνουμε μια πληρέστατη έκθεση που θα είναι χρήσιμη και για την Ουκρανία. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήμουν στην αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου που επεσκέφθη την Ουκρανία και μπορώ να σας πω ότι επέστρεψα με ανάμεικτα συναισθήματα. Είδαμε κάποιες διαμαρτυρίες, εκεί είδαμε πολλά προβλήματα και παρατυπίες, αλλά είδαμε και καλά σημάδια. Συμφωνώ με την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου όσον αφορά τη θητεία του Κοινοβουλίου, διότι έτσι αφαιρείται και ένα σημαντικό εμπόδιο της σταθερότητα. Ένα εκατομμύριο άνθρωποι βουλγαρικής καταγωγής κατοικούν στην Ουκρανία και νομίζω ότι είναι πρεσβευτές των, της ευρωπαϊκής ιδέας εκεί. Εντός του καθεστώτος θεωρήσεων διαβατηριών θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για εκείνους που έχουν αποσυνδεθεί από την, από την γη τους, γη τους εδώ και 300 χρόνια να ταξιδεύουν ελεύθερα στη χώρα τους και να εξαγάγουν τις ευρωπαϊκές ιδέες στην Ουκρανία. Ευχαριστώ κύριε Στογιάννοφ. επόμενος. Επόμενη μάλλον. Ευχαριστώ Πρόεδρο. Πρόσφατα η Ουκρανία γήτό ε, άλλων ανατολικών εταίρων. Ήταν στην πρώτη θέση ε, όσον αφορά την εφαρμογή των ευρωπαϊκών προδιαγραφών, των οικονομικών και νομικών μετατρο... μεταρρυθμίσεων κλπ. Οι πρόσφατες, τα πρόσφατα γεγονότα δημιούργησαν ε, κάποιες ανησυχίες λέει η κυρία Ανδρικιένε, και γι' αυτό πρέπει να εκφράσουμε τις ανησυχίες αυτές όσον αφορά τα άσχημα πράγματα που βλέπουμε και τις εξουσίες που δόθηκαν, παραδείγματος χάρη στις υπηρεσίες ασφαλείας, και τα μέτρα που λαμβάνουν αυτές οι υπηρεσίες ασφαλείας τρεφόμενοι κατά ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων και των μέσων ενημέρωση. Τούτο λεχθέντο πρέπει να πω και το εξή, ότι πρέπει να υποστηρίξουμε την ενταξιακή διαδικασία, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ε, θετικά κίνητρα ή αποτρεπτικά μέτρα. Ε, αλλά περισσότερο πρέπει να δώσουμε ένα δέλεαρ, θα έλεγα, καρότο. Θα πρέπει να φέρουμε πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση την Ουκρανία. Νομίζω ότι η ένταξή τη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στρατηγικό μα στόχο και θα πρέπει να βρούμε τα δειγμένα μέτρα για να φτάσουμε αυτό το στόχο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ανδρίκενα και ακολουθεί ο κύριος Μίλσκι. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, έχω μία ερώτηση μόνο προς όλους τους βουλευτές. Γιατί το χρειαζόμασταν σήμερα συγκεκριμένα αυτό το ψήφισμα για την Ουκρανία. Ε, Όντω, ε, πρέπει να βοηθήσουμε τη νέα κυβέρνηση, αλλά ποιο είναι ο πραγματικό στόχο μα, Θέλουμε να παρεύουμε πριν τι αυτοδιοικητικέ εκλογέ. Θέλουμε να επέμβουμε, ε, να μην αφήσουμε την Ουκρανία να ρυθμίσει η ίδια τα προβλήματά της. Στο αρχικό κείμενο λέγαμε ότι η κατάσταση είναι δεινή στην Ουκρανία γενικότερα. Δεν αληθεύει όμως αυτό. Θα έπρεπε να πηγεί το ψήφισμα την πραγματικότητα, τα πραγματικά γεγονότα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μίρσκι. Στο τέλος η κυρία Μπασέσκου. Κύριε, κύριε Πρόεδρε, μια πολύ σημαντική πτυχή της σημερινής συζήτησης ήταν η επικρίση σε σχέση με τη διαφάνεια και την αμεροληψία των τοπικών εκλογών που έλαβαν χώρα στις 31 Οκτώβρη. <clears throat> Υπήρξε πίεση από την κυβέρνηση στα μέσα ενημέρωσης και επίσης ο εκλογικός ε, νόμος δεν έδωσε πολλές ευκαιρίες στην αντιπολίτευση. Η Ουκρανία όμως παραμένει ένας πάρα πολύ σημαντικός εταίρος μας και εγώ χαιρετίζω τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαδικασία δημοκρατικοποίησης, κάτι που υπογραμμίστηκε και στη διάσκεψη κορυφής της Δευτέρας. Η εταιρική σχέση με την Ουκρανία είναι πάρα πολύ σημαντική και με την Ουκρανία, γιατί και οι δύο χώρες είναι πολύ σημαντικοί εταίροι στην περιοχή της μαύρη θάλασσα και σε ό,τι αφορά την ενεργειακή ε, αυτάρκεια ε, όπως και με τη Μολδαβία προβλέπεται να γίνει μια συμφωνία για συνοριακές δια... μετακινήσεις με την Ουκρανία όπως είχε γίνει και με τη Μολδαβία και η Ρουμανία έχει λοιπόν κάθε λόγο να μπορέσει να διευκολύνει την είσοδο των Ουκρανών στην Σοδαφό. ευχαριστώ πολύ. Για να κλείσει η συζήτηση τώρα δίνω το λόγο ε, στον <clears throat> κύριο Ντεχούχτ ο οποίος εκπροσωπεί την είπα το εκπρόσωπο κάτι Άστον. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα να απαντήσω στην ερώτηση που μου υπέβαλε η κυρία Βάλεαν για το, την νομοθεσία σχετικά με τις ε, δημόσιες ε, προμήθειες, τις αγορές. Ε, δεν ε, ασχολούμαστε με την επιότητα του νομοσχεδίου. Εμείς παρακολουθούμε τις έσχατες εξελίξεις ε, και για να στηρίξουμε ε, ε, οικονομικά τον ενεργειακό τομέα, η προϋπόθεση είναι να πληρούνται κάποια κριτήρια μέσα σε αυτή την νομοθεσία. Ε, Σχετικά με την ε, τωρινή κατάσταση στην Ουκρανία, η ανάλυση φυσικά πρέπει να γίνει και αυτό φαίνεται καθαρά στο ψήφισμα που θα ψηφιστεί αύριο. Πιστεύω ότι αν εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο ή μάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε να έχουμε κάποια επιρροή σε αυτό το θέμα, χρειαζόμαστε εγκάρσιες συμφωνίες σχετικά με το πώς ε, θα τοποθετηθούμε